Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, με συγχωρείτε, αλλά ε, για να προετοιμάσουμε τη συνεδρίαση χρειαστήκαμε περισσότερο χρόνο σαν συντονιστές για να ετοιμάσουμε την πολιτική συμφωνία την οποία επιτύχαμε και ελπίζω ότι έτσι θα ολοκληρώσουμε την εξέταση των τροπολογιών της Επιτροπής ε, Προπολογισμού και θα ολοκληρώσουμε όλα τα θέματα όπου υπάρχει πολιτική συμφωνία. Την επόμενη εβδομάδα θα χρειαστεί να ψηφίσουμε ορισμένα θέματα και θα σας πω στο τέλος συνεδριάσεως ποια θα είναι αυτά. Ξεκινώ λοιπόν με τις πιστώσεις ε, των εξωτερικών ε, υποθέσεων που είχαμε κρατήσει για το τέλος. μετά από μακρά συζήτηση μεταξύ των συντονιστών καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό βάσει της ε, δεύτερης εναλλακτικής λύσης, δηλαδή τον πίνακα ο οποίος μόλις ε, σας έδώσει. Αυτή είναι η βάση εργασίας ε, του, ε, συμβιβασμού. Αλλά θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουμε όλες τις γραμμές οι οποίες ε, αντικατοπτρίζουν την τελική συμβιβαστική λύση. Θέλω λοιπόν καταρχήν να σας παρουσιάσω την ε, πολιτική συμφωνία και εάν συμφωνήσετε την πολιτική συμφωνία και την υπερψηφίσετε τότε θα ψηφίσουμε ε, όλες τις γραμμές οι οποίες βρίσκονται στο, στη δεύτερη εναλλακτική λύση ε, εκτός από την ε, τελική συμβιβαστική λύση όπου για τεχνικούς λόγους θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να ε, εξετάσουμε σε 5-6 γραμμές το ακριβές ποσό και να τα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Θέλω επίσης να σας προτείνω να ψηφίσουμε συνολικά σαν μια ομάδα ε, όλες ε, τις, όλα την κατηγορία 4. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις. Ας παρουσιάσω την ε, πολιτική συμβιβαστική λύση και ο εισηγητής θα παρουσιάσει τα σχόλιά του αν επιθυμεί. Το πρόβλημα ήταν το εξής. Έχουμε μία πολιτική συμφωνία μεταξύ των ομάδων για να μην υπερβούμε στην κατηγορία 4 όπως άλλωστε και σε άλλες κατηγορίες ε, το, την οροφή των ε, δημοσιονομικών προοπτικών. Όλες οι τροπολογίες ε, τις οποίες εξετάσαμε μέχρι τώρα οδηγούσαν σε μία υπέρβαση περίπου 41,5 εκατομμυρίων, δηλαδή πάνω από 40 εκατομμύρια, υπέρβαση του, ε, ε, της οροφής και έπρεπε να βρούμε 41,5 εκατομμύρια. Η πολιτική συμφωνία στην οποία καταλήξαμε ε, συνίσταται στο να πούμε ότι θα κάνουμε αντίστοιχες εξοικονομήσεις κατανέμοντας 50-50 περίπου τα μέτρα, τα συνοδευτικά της συμφωνίας για την μπανάνα και τη γραμμή ICI+. Plus, δηλαδή ε, συνεργασία με τις βιομηχανοποιημένες χώρες. Αυτή είναι η πολιτική συμβαστική λύση στην οποία κατέληξε η Επιτροπή ε, Προϋπολογισμού. Η ε, επιλογή των γραμμών αυτών οφείλεται και πρέπει να το πω δημοσίως, άπαξ και τώρα μας παρακολουθεί το κοινό, όχι διότι δεν ενδιαφερόμαστε ή αντιτιθέμεθα ή στην ε, συμφωνία η οποία έγινε ε, από την Ευρώπη με τις ε, χώρες που παράγουν μπανάνες ή με τις χώρες ICI συν αλλά θεωρήθηκε αναγκαία για να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαιρετίζω τον Γενικό Διευθυντή και στο Συμβούλιο για να αντιληφθούν ότι άπαξ και το Συμβούλιο αρνείται να ε, εξετάσει ε, την ε, αύξηση της οροφής ορισμένες κατηγορίες του κεφαλαίου 4 θα χρειαστεί να υπάρξουν θυσίες πολιτικές Κατά τις τρεις αυτές ημέρες έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για να ε, μπορέσουμε να παραμείνουμε κάτω από τις οροφές. Επί 15 χρόνια ε, συνήθως ε, ψηφίζαμε τροπολογίες πέραν της οροφής. Αυτή τη φορά όμως δεχθήκαμε να περιοριστούμε αλλά και το Συμβούλιο πρέπει να αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό και από πλευράς ε, των ε, Υπουργών ε, Οικονομικών δεν θα πρέπει να ακούμε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν κάνει τίποτα, δεν εξυπηρετεί τίποτα και πρέπει να τον περιορίσουμε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι οι επίσημες δηλώσεις που γίνονται στον ΟΗΕ δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Λοιπόν, βάσει αυτής της αρχής Δηλαδή να βρούμε 41,5 εκατομμύρια είναι μια τάξη γέθους υπό επιφύλαξη της τεχνικής επαλήθευσης μεταξύ των δύο αυτών γραμμών με αυτή την επιφύλαξη θα υποβάλω την συμφωνία εις, ε, το, ε, για ψήφιση. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ένας κατά. Αποχές. Δύο αποχές. Ευχαριστώ. Αυτή η ανάταση χειρών μπροστά ε, στα μέσα ενημέρωσης ε, τα ε, που είναι διεθνή είναι πολύ σημαντική κίνηση. Οπότε τώρα ψηφίζουμε ομαδικά τον πίνακα της δεύτερης αναλλακτικής λύσης μείον τις γραμμές δεν είχαμε χρόνο να τις ε, διαγράψουμε ε, τις γραμμές της μπανάνας και του ICI συν. Κατά. Τέσσερις. Αποχές. Δεν έχουμε αποχές. Οπότε και η δεύτερη εναλλακτική λύση ε, έχει εγκριθεί. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στις, ε, ε, στις παρατηρήσεις. Έχουμε ε, ένα σύνολο παρατηρήσεων και θα ήθελα να είμαι βέβαιος ότι έχετε το σωστό έγγραφο που ονομάζεται 4RAP προτάσεις των συντονιστών στις σελίδες 13 και 14. Alors attendez. Euh, on, on, on achève de distribuer. Est-ce que, est que je peux commencer Βλέπω ότι κατανείμεται. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ε, δεν είναι ένα νέο έγγραφο, είχε δοθεί την ε, Δευτέρα και απλώς υπάρχει ε, μία, ένας προφορικός συμβιβασμός που θα παρουσιάσει η συγγήτρια. Λοιπόν, ε, ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία 384 τη Ρέτζι. Κατά. Δύο κατά. Εγκρίνεται. Στο 4662 του κυρίου Έρενχάουζερ ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46-49 ε, ε, του κυρίου Έρενχάουζερ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Έχουμε την 494, μία οριζόντια, μία οριζόντια α, ε, ψηφοφορία ποιος είναι υπέρ. Η συγγήτρια είναι υπέρ αλλά πρέπει να κάνουμε ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Και εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω. Ξεκίνησε η ψηφοφορία, εγώ δεν ψηφίζω. Ψήφισε και η Αντιπρόεδρος. Ωραία. Λίγη ψηφοφορία. 18 υπέρ, 21 κατά. Άρα απορρίπτεται. Η 368 της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ποιος είναι ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42-40 του κυρίου ή της κυρίας Τόγια και άλλων. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Οι σοσιαλιστές είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Όλοι οι υπόλοιποι. Βλέπω ότι είναι τραγικά απομονωμένοι σοσιαλιστές και η τροπολογία αποσύρεται. Οι 342 και οι 722 ποιος είναι υπέρ. Αποχές εγκρίνονται. 846 της ΓΟΕ. Ποιος είναι υπέρ. Η συγκήτρια είναι κατά. Ποιος είναι κατά. Όλοι οι υπόλοιποι. Λυπάμαι αλλά απερίφθη. Μετά έχουμε την 343 ε, η εισηγήτρια είναι υπέρ, κατά, αποχές, μία αποχή και εγκρίνεται. Πολλές τροπολογίες ε, στην 344 ποιος είναι υπέρ, κατά. Και η Μπάρμπαρα είναι κατά. Ε, αποχές, μία αποχή εγκρίνεται. Η 334 της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ε, ε αποχές εγκρίνεται. Η 354 είναι σχόλια της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο εισηγητής είναι ε, υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. Η 594 των πρασίνων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται εφόσον τα μεγάλα κόμματα αντιτίθενται. Η 345 της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ε, απορρίπτεται. Α, με συγχωρείτε. Η 390 ποιος είναι υπέρ. Για τις μπανάνες. Κατά. Αλλά εγκρίνεται γιατί υπερισχύει η κεντροδεξιά. 364 της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Κατά. Αποχές. Η 595 των Πρασίνων. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η 333 της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην ίδια γραμμή υπάρχουν πολλές τροπολογίες. Η 4214 του κυρίου Γκαρίγκα και της κυρίας Γκρέσλε που είναι οριζόντια τροπολογία που θα επανέλθει. Ο συγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Η φιλελεύθερη. Εγκρίνεται. Η 369 της τροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, ο εισηγητής είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Δύο αποχές. Η 642 ε, του κυρίου Χόγκλουντ και των φιλελευθέρων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Η συγγήτρια και ο James Έλλες είναι αντίθετοι. Αποδεικνύονται ορισμένα πράγματα. 483. Ποια είναι η άποψη του συγγήτρες. Είναι τροπολογία Έλλης. Κατά. Αποχές. Δύο αποχές. Εγκρίνεται. 585 των πρασίνων. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν ψηφίζω. Λίγοι. Οι 23 υπέρ, 17 κατά εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 16 ε, των σοσιαλιστών και της Επιτροπής Αναπτύξεως. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 365. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41-92 του Λάσλο Σούριαν. Η συγκίτρια είναι κατά. Κατά. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Είμαστε 42 παρόντες. Ψηφίζουμε όλοι. Λίγη η συζήτηση. 22 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42. Της δικής μας επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Αποχές δύο εποχές Στις 43 της ίδιας επιτροπής, εισηγήτρια υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 495 καλύπτεται. 20 της Επιτροπής Ανάπτυξης υπέρ, κατά, αποχές, 23 de la même commission du développement, le rapporteur est toujours pour. Super. κατά, αποχές, εγκρίνονται. 32 της Επιτροπής Ανάπτυξης. Με συμφωνία της ηγετίας υπέρ, κατά, αποχές. Adopté. Εγκρίνεται. Le 45 de Monsieur Mitchell. Η Μίτσελ. συγκίτρια είναι κατά. Υπέρ. Το ΕΛΚ κατά. Η μη, Και η συγκίτρια φυσικά. Η συγκίτρια δεν είναι ΕΛΚ. Η, συγκίτρια δεν έχει φίλο πολιτικά φίλο Το ξέρω, ξέρω γιατί μιλάω, γιατί έχω υπάρξει και εγώ εισηγητή. Απορρίπτεται λοιπόν. 22. Επιτροπής Ανάπτυξης. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην 31 υπάρχει μια συμβαστική τροπολογία. Όντως, καταλήξαμε σε μια συμφωνία για το κείμενο. Σας ε, μοιράστηκε με email αλλά έγινε άλλη μία αλλαγή. Και επανέρχεται το αρχικό κείμενο των σοσιαλιστών, σας το διαβάζω. Τμήμα αυτών των πιστώσεων θα μπει στο αποθεματικό μέχρι ότου η Κομισιόν η υποβάλλει μια, ένα έγγραφο πολιτικής δεσμευτικό που λέω ότι το πακέτο για το κλίμα είναι όντως προσθετικό. Δηλαδή να δίνουμε πόρες ένεργες σε εταίρους με ένα γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο και δεν θα είναι σε βάρος προγραμμάτων συνεργασίας και ανάπτυξης όπως και παρουσίαση των οικονομικών εισφορών των κρατών μελών στον Μηχανισμό Ταχείας Παρέμβασης με βάση τα κριτήρια των δικαιούχων και συμφωνίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θέλετε να συνεχίσω? Πρόεδρος, όχι, όχι σε σχέση με το γραπτό κείμενο αποκαθιστούμε τη φράση που είχε διαγραφεί πριν. Συνεχίζεται. Το υπόλοιπο έχει μοιραστεί. Η πρότασή μου είναι να ψηφίσουμε υπέρ. Έλεγα. Όχι. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 708 καλύπτεται. Υγεία. 644. Φιλελεύθερον κύριος Άλβαρο. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43-42. Η, η είναι υπέρ. Υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. 18 υπέρ, 20 κατά απορρίπτεται. 594 υπέρ 593 ε, κατά προσοχές, η συγγήτρια και η κυρία Αντιάσεν εγκρίνεται η ευρωπαϊκή πολιτική είναι πάρα πολύ σύνθετο πράγμα 355 de la Commission des Affaires étrangères. Le rapporteur est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 probablement la semaine prochaine, et je l'espère en bloc, les commentaires. Voilà où nous en sommes. Donc Sidonia est prête, je lui donne la parole. Eh, eh, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους σας για την συνεισφορά σας. Θα τα πάρετε αυτά. Ζητώ συγγνώμη εξ ονόματός μου και της γραμματείας. Αλλά συμφωνήσαμε μόλις χθες το βράδυ για αυτά. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό στο ρεύμα στο τμήμα του κτηρίου όπου εργαζόταν η γραμματεία. Και αυτό επεξηγεί την καθυστέρηση, το πρόβλημα με την επικαιροποίηση του πίνακα. Παρ' όλα αυτά έχω κάποια σημαντικά μηνύματα που μπορώ να σας δώσω άμεσα τώρα. Πάνω από 150 προγράμματα πετύχαμε από πλευρά τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Επιτροπή Προπολογισμών. Αυτό που κάναμε σχετικά με τον Ιούνιο ήταν κάποια καινοτομία τα όσα έσυλαν τα μέλη στάθηκαν προς αναθεώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σαν ένας τρόπος να εξεταστούν κάποιες ιδέες, διότι οι προκαταρκτικές δράσεις, σύμφωνα με τη δική μας ερμηνεία, είναι τμήμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που θα προέλθει νομοθετικά και πρέπει να είναι πραγματικά καινοτόμος και καινούρια. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξετάσουμε και να ελέγξουμε και ήταν επικοδομητική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό να δούμε σε σχέση με τα προηγούμενα ή σημερινά προγράμματα να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις ιδέες. Είμαστε σίγουρα καινοτόμοι και όχι επαναληπτικοί. Αυτό λοιπόν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστούμε για τη συνεργασία που ήταν ομαλή, επικοδομητική. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι κάποια εντολή για μας, εντάξει, προφανώς. Είναι μια σύσταση για αξιολόγηση. Εν τέλει όμως τελικά δεν είναι κάποια δεσμευτική αξιολόγηση. Επίσης και κάποιες αψυχινοβουλευτικές επιτροπές και οι Ευρω... κάποιοι ευρωβουλευτές δεν ήταν σε θέση να έχουν έτοιμα τα προγράμματά τους, τα σχέδιά τους τον Ιούνιο και έτσι δεν μπορούσαν να αξιολογηθούν αυτά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Είμαι εντυπωσιασμένη από την δημιουργικότητα των μελών και είναι μια πρόκληση για μένα αυτή η δημιουργικότητα συναδέφου, συναδέφων και ε, βλέποντας τις, ε, τα πιλωτικά προγράμματα και τις προκαταρκτικές δράσεις είναι μία διάβαση, ένα ταξίδι μέσα από την δημιουργικότητα του σώματος με πάσης φύσεως ε, εγχειρήματα και προγράμματα για την επιλογή, πολύ δύσκολη υπόθεση για μένα ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν να δώσω κονδύλια, πόρους στα εξελισσόμενα υποεξέλιξη προγράμματα προκατακτικών δράσεων και πιλωτικών. Δεν ξεκινάμε νέα πράγματα, αλλά αντίθετα διασφαλίζουμε ότι κάποια επιτυχή προγράμματα που βρίσκονται υποεξέλιξη θα διασφαλίσουν τη χρηματοδότησή τους για τα επόμενα χρόνια. Κάποια από τα προγράμματα είναι ήδη υφιστάμενα που διασφαλίζουν κονδύλια για να συνεχιστούν στο μέλλον. Από κοινού, εγώ και οι συντονιστές προσπαθούσαμε να βρούμε ένα συμβιβασμό. Συμβιβασμό που θα δίνει, διακόπτει θα δίνει το πράσινο φως ή μια δυνατότητα στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές και διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες αλλά ήταν δύσκολη η ισορροπία που έπρεπε να επιτευχθεί. Πιστεύω επίσης ότι οι αποκαλούμενες μικρότερες ομάδες μικρότερες κοινοβουλευτικές ομάδες πρέπει να έχουν και εκείνες κάποια προγράμματα. Γιατί αν ψηφίσουμε αριθμητικά μπορεί να καταψηφιστούν. Δεν πρέπει όμως να μην έχουν τίποτα. Πρέπει και οι μικρότερες ομάδες να έχουν κάποια πιλωτικά προγράμματα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν θέματα που έχουν λιγότερο, ας το πω έτσι, ληφθεί υπόψη. Τώρα, σημαντικό είναι να δούμε για την κατανομή μεταξύ των κεφαλαίων των κατηγοριών. Να δώσω κάποια επεξήγηση τι έγινε. Περιοριζόμαστε από το πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας στα όρια της, που περιορίζει τα συνολικά πλαίσια για πιλωτικές δράσεις και προκατακτικά σχέδια. Ήταν ένας από τους περιορισμούς, αλλά δεν είχαμε πρόβλημα, γιατί δεν φτάσαμε στα όρια, δεν είχαμε καν κονδύλια ούτως ή άλλως ε, πόρους στο περιθώριο. Γι' αυτό τα περιθώρια στις κατηγορίες ήταν τα όρια μας περισσότερο αυτά παρά η διοργανική συμφωνία. Έτσι λοιπόν, εν τέλει, αυτό που έγινε ήταν ότι περισσότερα, τα περισσότερα προγράμματα που είχαν κατατεθεί όσον αφορά την κατηγορία 1α δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει σε σχέση με την καινοτομία, την, την επιχειρηματικότητα κτλ. Και για την κατηγορία 1β όχι τόσα πολλά και αρκετά στην κατηγορία 2, πράγμα που δείχνει τώρα ότι στην Γεωργία και στην Αλία οι ευρωβουλευτές χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις δράσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Τώρα, στον κατάλογο που ελπίζω ότι θα έχετε στα χέρια σας τώρα, ναι, ναι, τον έχετε, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, σε αυτόν τον κατάλογο υπάρχουν δύο σφάλματα που αμέσως πρέπει να σας επισημάνω. Και αυτά είναι ως εξή. Στην πρώτη σελίδα, στην 150231 γραμμή, το ποσό είναι λάθος, δεν είναι 2,4 εκατομμύρια, είναι 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Αντί να περιμένουμε λοιπόν να έχουμε ένα νέο αντίτυπο, να πάρετε τα μολύβια σας και να διορθώσετε αυτό το ποσό. Αντί 2,4 εκατομμύρια είναι 1,4 εκατομμύρια αυτή η γραμμή στο 150231. Και μετά από αυτά που είπα πιο πριν και αυτά που συμφωνήθηκαν από τους συντονιστές, πραγματικά προστίθεται στην κατηγορία 4, κάτι το οποίο δεν έχετε στους καταλόγους σας, στον κατάλογο μέχρι τώρα, θέλω να το να προσθεθεί και θέλω την υποστήριξή σας σε αυτό το σχέδιο να προσθεθεί πιλωτικό πρόγραμμα της ομάδας Ενωτικής Αριστεράς της ΓΟΕ για τα στην κατηγορία 4. Το ποσό είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι το πακέτο που προτείνω συνολικά να, χρησ... να εγκριθεί από πλευρά σας. Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, αν βρείτε κάποια άλλα λάθη, έχετε κάποια σχόλια, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολλοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο και αμέσως θα τους το δώσω. Θα ήθελα να είμαι βέβαιος ότι όλοι έχουν αντιληφθεί πλήρως τις δύο διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στην προτελευταία έκδοση του ε, πίνακα που είναι σωστή. Δηλαδή με την ε, τροπολογία της Γκούε ενώ ο πίνακας ε, του Προέδρου και του εισηγητή έχουν δύο λάθη. Στην πρώτη σελίδα το Power Cost and Studies from EMP είναι επιπλέον 1,4 εκατομμύρια και όχι 2 και στη σελίδα 2 πρέπει να προσθέσουμε ε, ένα πιλωτικό πρόγραμμα της ΓΚΟΕ για τα θύματα των βασανισμών, άλλο ένα εκατομμύριο. Πρέπει λοιπόν να ε, γίνει αυτή η διόρθωση. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω για τα νέα μέλη είναι ότι όπως το είπε ο εισηγητής, η συγγητρία Γνωρίζετε όλοι ότι έχουμε ένα, μια οροφή κατά κατηγορία δαπανών 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1 β, 2, 2 β και το καθεξής. Έχουμε όμως και ένα συγκεκριμένο πλαφόν για τις ε, πιλωτικές ενέργειες και όπως είπε η συγκήτρια δεν υπερβαίνουμε αυτή την οροφή γιατί δεσμευόμαστε από τους οροφές των πέντε κατηγοριών. Οπότε ο ευρωπαϊκός ε, προϋπολογισμός για το Κοινοβούλιο είναι πολύ περιοριστικός. Είμαστε δεμένοι με ζωρολομανδία κατά κάποιο τρόπο. Δεν μπορούμε να κουνηθούμε δηλαδή. Από την άλλη μεριά το είπε και το ξαναλέω και εγώ. Θα ψηφίσουμε τα ποσά, όχι τα σχόλια, ξέροντας ότι ορισμένοι συνάδελφοι μπορεί να θέσουν ερωτήσεις, ορισμένες προτάσεις για πλωτικά προγράμματα που υπέβαλαν δεν επιλέγησαν ως επιλωτικά προγράμματα προτείνουμε να ληφθούν υπόψη στα σχόλια για τις τακτικές γραμμές του προπολογισμού που ψηφίστηκαν χθες και προχθές. Φυσικά αν υπάρχουν ερωτήσεις, η συγγήτρια θα απαντήσει. Αν Γένσεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ επίσης την εισηγήτριά μας που είχε τεράστιες δυσκολίες να καλύψει αυτή τη δουλειά και έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά προσπαθώντας να καταλήξει σε ένα συμβιβασμό. Νομίζω σε σχέση με αυτή τη δημοσιονομική διαδικασία μας έμαθε αυτή ότι υπάρχουν πραγματικά πολλές καλές ιδέες, καινοτόμες, επινοητικές ιδέες στο, στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά ότι επίσης πρέπει να συμπτύξουμε τις διαδικασίες μας ε, για να είναι δυνατόν οι μελλοντικοί εισηγητές να έχουν ευκολότερο βίο και πιο εύκολα να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Πρέπει να συμπτύξουμε, να κάνουμε πιο αποτελεσματικούς τους κανόνες του παιχνιδιού, ώστε να διασφαλίσουμε να εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Ξεκίνησε η Utah Χάουγκ όταν ήταν εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό με αυτό. Και κάθε χρόνο κάνουμε αυτή την προσπάθεια και πρέπει να το καταφέρουμε στο τέλος και να γίνουμε, όλο και καλύτεροι. Έχω κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά τον νέο κατάλογο. Μία ερώτηση. Υπήρχε στο παρελθόν κάποια παρατήρηση σε σχέση με το 04 για την πρόληψη της κατάχρησης και της βίας των βασανιστήριων. Θα ήθελα να ρωτήσω την εισηγήτρια τι γίνεται σχετικά, διότι το ανέφερε προγράμματα που ε, βρίσκονται υπό εξέλιξη και θα εκπνεύσουν δεν μπορούν να αλλάξουν την τελευταία στιγμή, στην τελευταία φάση. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνέχειά τους. Αυτός θα πρέπει να είναι ο λόγος. Έτσι εντάξει. Τώρα και για το ε, ποσό που θα ήθελα και θα με ευχαριστούσε να αυξηθεί το 1,4 εκατομμύριο είναι, δεν είναι καλός όμως, είναι εντάξει. Έχω κάποια ερώτηση σχετικά όμως με τα εξωτερικά θέματα, εξωτερικές υποθέσεις, foreign affairs, την τροπολογία 363 στην, στο γραμ, στην γραμμή 190406 κοινωνία των πολιτών ΕΕ Ρωσία πρόταση να διαγραφεί μια φράση στα σχόλια στις παρατηρήσεις. Θα θέλαμε από την ομάδα Άλτε να γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία για αυτή τη διαγραφή. Δεν συμφωνούμε με αυτή τη διαγραφή. Θεωρούμε ότι αυτή η παρατήρηση, αυτό το σχόλιο είναι σημαντικό. Και επειδή είναι ένας τρόπος, είναι έτσι διοργανωμένο αυτό που είναι σημαντικό αυτό το σχόλιο μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και το τελευταίο Μπορούμε να υποστηρίξουμε την τροπολογία της ΓΚΟΕ για τα βασανιστήρια, παρότι δεν βρίσκεται στο, για τα θύματα βασανιστήριων, παρότι δεν είναι στον κατάλογο, αλλά ήθελα να ζητήσω κάτι. Με την τροπολογία των πρασίνων που γίνεται λόγος για να ενταχθεί στην κατηγορία 5 για το EEAS, τι έγινε με αυτή την τροπολογία, μπορείτε να μου πείτε. Αυτές είναι οι κυριότερες παρατηρήσεις και ερωτήσεις μου. Κατά τα άλλα θα έλεγα ότι η ομάδα Άλντε είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με αυτά που έχουν επιτευχθεί και έχουν προταθεί. Είναι νομίζω ένα σωστό συμβιβασμό και μπορούμε να τον υποστηρίξουμε. Merci. Merci beaucoup, Anne. Σας ευχαριστώ πολύ, Αν. Η συγγύτρια θα απαντήσει στις παρατηρήσεις. Δαμιάν Αμπάντ. Oui, merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ συγχαίρω την εισηγήτρια και το εξαιρετικό της έργο και το συμβασμό που πετύχαμε. Τονίζω μόνο, επειδή είμαι νέο μέλος, όπως και άλλοι συνάδελφοι, είναι αρκετά περίπλοκο. Περίπλοκη σαν διαδικασία. Αν είμαστε λιγότερο αδιαφανείς, θα ήταν καλύτερα. Οι συντονιστές, ο ρόλος τους είναι επιφανής θα έλεγα. Καλό θα είναι όμως όλοι μαζί να συνεργαζόμαστε για να καταλάβουμε τους μηχανισμούς για τα πιλωτικά προγράμματα ή θα αποφασίσουμε ότι θα τα υποστηρίξει η ομάδα οπότε από την αρχή της διαδικασίας θα πούμε ότι οι ομάδες προτείνουν τα πιλωτικά προγράμματα ή αλλιώς θα επιτρέψουμε επιμέρους αιτήματα πιλωτικών προγραμμάτων μερικά από τα προγράμματα όπως αυτά τα αξιολόγησε η Κομισιόν και μετά δεν επελέγησαν. Μεθοδολογική παρατήρηση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δυσκολίες στη διαπραγμάτευση, αλλά θα έπρεπε νομίζω στο μέλλον να υπάρχει αυτή η στενή συνεργασία με όλα τα μέλη. Για να έχουμε βελτίωση όσον αφορά την παρουσίαση των προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε αγαπητέ συνάδελφε. Χέλγα. Uh, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σιδονία για τη δουλειά που έκανε στην εξέβρεση συμβιβασμού. Θα θέλω να επανέλθω όμως στο ήδη προαναφερθέν θέμα από την Άννα για την υποστήριξη διαμεσολάβηση στην EAAS και δεν το βρίσκω εδώ σε αυτό το συμβιβασμό και γι' αυτό δεν θεωρώ ότι με ικανοποιεί και πρέπει αυτό να καλυφθεί. Ευχαριστώ. Merci. Θα είμαι πολύ σύντομος συμφωνώ με τους άλλους και προσθέτω τη φωνή μου στις ευχαριστίες για την εισηγήτρια. Έκανε πραγματική προσπάθεια να ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες. Φυσικά δεν είναι δυνατόν όλες οι επιθυμίες να ικανοποιούνται πάντα, αλλά είναι μια σωστή θα έλεγα πρόταση αυτή. Θέλουμε να έχουμε κάποιες ξεχωριστές ψηφοφορίες στα σχόλια στις παρατηρήσεις, αλλά θα επανέλθουμε όταν έρθει η ώρα. Ευχαριστώ, αυτά είχα να πω. Ε, personne Εκ μέρους του ΕΛΚ κανένας δεν μίλησε. Ο κύριος Λαβία. Δεν μιλώ εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ως μέλος της Επιτροπής Προπολογισμών θα μιλήσω. Ευχαριστώ και εγώ τη Συντόνια για τη δουλειά της. Προσωπικά βέβαια δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένο γιατί έγινε μια μικρή αυλεψία. Ένα πρόγραμμα για την αμοιοτροφική ε, σκλήρωση, σκλήρινση, συγγνώμη, δυστυχώς δεν επελέγει. Βέβαια στη γραμμή του προπολογισμού προβλέπεται προτεραιότητα για την πολλαπλή σκλήρινση. Είναι δύο διαφορετικές γενετικές ασθένειες, διαφορετικές. δεν δράσαμε σωστά. Δημιουργήθηκε σύγχυση εκ μέρους μας μεταξύ δύο διαφορετικών γενετικών ασθενειών. Στις, ή στις παρατηρήσεις θα καλυφθεί και η αμοιοτροφική σκλήρινση ή θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να επαναεισαγωγή στο αιτήματο. Πρόεδρος. Επιτέλους και ένας επίσημος εκπρόσωπος του κόμματος για να αποσαφινιστεί η κατάσταση. Βλέπω ότι η γνωμοδότηση του ΕΛΚ εκφράστηκε από την εισηγήτρια που κάποτε ανήκε στη δική μας ομάδα και θα ανήκει στο μέλλον πάλι ξανά σε μας. Μάλιστα, λοιπόν, επιτρέψτε μου απλά να πω ότι για την μειοτροφική πλευρική ε, σκλήρωση, αυτά που ακούσαμε τον Τζοβάνι, ότι ήταν ένα από τα θέματα των τελικών εξετάσεών μου κατά τις ιατρικές μου σπουδές και ακολουθώ απόλυτα τον Τζοβάνι στην πρότασή του. Ευχαριστώ. Merci. Jutta και η Jutta τώρα. Σας ευχαριστώ. Κάπως θα έλεγα και εγώ φταίω για το ότι εχθές όταν είχαμε συμφωνήσει όσον αφορά τον κατάλογο των πιλωτικών σχεδίων ότι αυτό δεν εντάχθηκε. Και για ακριβώς αυτόν τον λόγο και το ομολογώ ότι σκέφτηκα ότι έχουμε τώρα σχόλια για τη σκλήρωση. Ε, λοιπόν, δεν χρειάζεται επιπρόσθετα να έχουμε ένα πιλωτικό σχέδιο που θα εντάξουμε. Μια και όμως Ούτως ή άλλως την επόμενη εβδομάδα τα πιλωτικά προγράμματα τα οποία δεν εντάχθηκαν αλλά όπου βλέπουμε ότι μπορούν να ενταχθούν στις παρατηρήσεις και στα σχόλια που ούτως ή άλλως θα πρέπει να ψηφίσουμε. Είμαι υπέρ και με, αυτό, με αυτή τη δεύτερη μορφή σκληρώσεως να την εντάξουμε στα σχόλια, στις παρατηρήσεις, ώστε και οι δύο να καλύπτονται. Και θα έλεγα με αυτόν τον τρόπο σωστά θα μπορέσει να διασφαλιστεί και να ενταχθεί έτσι. Κύριε Σχάρτον, κύριε Πρόεδρε, πιθανότατα δεν θα επηρεάσει πλέον την ε, στάση στην ψηφοφορία και το πώς θα ψηφίσουν οι συνάδελφοι, αλλά στα πρακτικά παρακαλώ να καταχωρηθεί το εξή. Δεν υποβάλλω κάποια πρόταση εδώ που από τα μέλη έχει υποβληθεί και γι' αυτό δεν ξέρω αν αυτή είναι και η σωστή προσέγγιση. Για να απαντήσω στον κύριο όπως είπε η Αν Γένσεν, και εγώ θεωρώ και συμφώνησαν οι συντονιστές χθες πρέπει να έχουμε μια πιο αυστηρή ε, μέθοδο εργασίας για να διευκολυθούν αυτά τα πιλωτικά προγράμματα γιατί το θέμα είναι πολύπλοκο και λεφτά πολλά δεν υπάρχουν αυτό ισχύει για όλες τις κατηγορίες οι αρμόδιες επιτροπές μας παίζουν το ρόλο τους κάνοντας προτάσεις οι ομάδες επίσης Ο κάθε βουλευτής μπορεί να κάνει πρόταση και πρέπει και τα προγράμματα να είναι ρεαλιστικά. Σας διαβεβαιώνω ότι του χρόνου η διαδικασία θα είναι πιο σαφής, πιο αποτελεσματική, τηρώντας τις αυστηρές προθεσμίες που έχουμε. έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να ε, υποβάλει και να υποστηρίξει το πρόγραμμά του. Η συγγήτρια τώρα θα δώσει απαντήσεις. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ όλους. Και σε σχέση με εκείνα που αφορούσαν το να βρεθούν κάποια στοιχεία που λείπουν στον κατάλογο. Γι' αυτό το πρόγραμμα των Πρασίνων για τη διαμεσολάβηση στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λείπει για 600.000 ευρώ δεν εντάχθηκε επειδή είχαμε συζήτηση γιατί αν θα έπρεπε να ενταχθεί στα, στις παρατηρήσεις ή όχι θα επανέλθουμε λοιπόν στην αρχική δέσμευση να συμπεριληφθεί αυτό το πρόγραμμα στην κατηγορία 5 εκεί θα προσθεθεί στον κατάλογο 600.000 ευρώ πιστώσεις υποχρεώσεων Συντόνια, συγγνώμη προτείνεις να προσθέσουμε μία γραμμή. Δηλαδή, να πάρουμε το πρόγραμμα των πρασίνων που δεν υπάρχει πια, επειδή έχουμε περιθώριο στην κατηγορία αυτή. Ακριβώς όπως το εξηγείτε και είχε συμφωνηθεί χθε στους συντονιστές λόγω του blackout του βραδιά της και τα λοιπά δεν προσθέθηκε σε αυτόν τον κατάλογο. Και θα έπρεπε να το είχα αναφέρει αλλά δεν το έκανα. θα, θα έπρεπε να είχε ενταχθεί αλλά δεν εντάχθηκε. Όταν δεν υπάρχει ηλεκτρισμός ξεφανίζονται οι τροπολογίες των πρασίνων. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι πολιτικά ορθό για τους πρασίνους. Uh, Ένα άλλο θέμα το οποίο είχε αναφερθεί αν δεν κάνω λάθος, από την κυρία Γένσεν για κάτι το οποίο ανήγγυλα εχθές και θα επαναλάβω, που συσχετίζεται σε τροπολογίες που αλλάζουν παρατηρήσεις σε υφιστάμενα προγράμματα και προκατακτικές δράσεις. Δεν μπορώ να συστήσω να υπερψηφιστεί. Γιατί? Διότι καταρχήν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για παρατηρήσεις σε πληρωμές μόνο. Λοιπόν, όταν θα έχουμε το προϋπολογισμό και θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου, δεν υπάρχει δυνατότητα πλέον για άλλε θέσει. Έτσι λοιπόν είναι ανεδαφικό να αλλάξουμε τα σχόλια όταν έχουμε μόνο πληρωμές για συμβάσεις που έχουν ήδη συναυθεί και υπογραφεί. Κατανοώ για τις αλλαγές αυτές, αλλά θα είναι κάποια κίνηση σε σχέση με τους συντάκτες. Όμως είναι ανεδαφικό, είναι ξεπερασμένο πλέον αυτό σε αυτή τη φάση. Είναι υπερβολικά αργά πολύ καθυστερημένο να γίνει κάτι τέτοιο αλλαγή. Έχουν ξεκινήσει αυτά τα προγράμματα, βρίσκονται υπό εξέλιξη με συμβάσεις και δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Υπήρξε, υπάρχει καθυστέρηση. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να γίνει αυτή η αλλαγή σε σχέση με την πρόταση. Ένα άλλο θέμα. Έχω κάτι άλλο ακόμα. Μια άλλη παρατήρηση εδώ. Ποια είναι, μια στιγμή. Γενικά για τις παρατηρήσεις. Εδώ έχουμε δύο πράγματα, δύο θέματα. Ένα θέμα συνδέεται με τις παρατηρήσεις επί των προτάσεων που δεν έχουν ενταχθεί στον κατάλογο που όμως θα μπορούσαν να προσθεθούν σε κάποιες παρατηρήσεις κονδυλίων για τα τόσα άλλα πιλωτικά προγράμματα. Είναι πολύ δουλειά να δούμε τις παρατηρήσεις, τι θα γίνει αν θα ενταχθούν στο υφιστάμενο κονδύλιο ή όχι. Θα πάρετε ένα φυλάδιο με όλες αυτές τις προτάσεις ε, για αυτά τα σχόλια και παρατηρήσεις, για τα κονδύλια, για την ψήφιση την Δευτέρα. Θα τα πάρετε έγκαιρα, εκ προημίου, ώστε να μπορέσετε να δείτε τι γίνεται σε σχέση με αυτά τα σχόλια. Ένα άλλο θέμα είναι οι παρατηρήσεις που συνδέονται με τις πιλωτικές δάσεις και προκατακτικές δάσεις που έχουμε επί ως πρόταση. Θα πρότεινα πάλι να υπάρξει ένας κατάλογος αυτών. Καταρχήν, οι παρατηρήσεις αυτές που αρχικά συνδεόντουσαν με τα αρχικά προγράμματα και πιλωτικές δράσεις και τις τροπολογίες, όμως σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε συγχωνεύσει, έχουμε συνδυάσει. Γι' αυτό πρέπει να δούμε τα κείμενα, πώς συνδυάζονται με αυτή τη συγχώνευση για τις παρατηρήσεις. Και κατά κάποιο τρόπο πολλές φορές είναι τροπολογίες που πρέπει ξεχωριστά να ψηφιστούν διότι δεν ξέραμε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα όλων αυτών των διαπραγματεύσεων και πώς θα επηρέαζε το ποσό. Για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο θέτει ο Τζοβάνι Λαβία για τη σκλήρωση, ανακαλύπτω την άγνοιά μου, πόσο μεγάλη είναι. Μελετώντας πιλωτικά προγράμματα και υποκατακτικές δράσεις και ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι είμαι για την ιατρική, θα μπορούσα να είχα κάνει λάθο κι εγώ και ίσω έπεσε και στην ίδια παγίδα η Γιούτα όπω και εγώ. Είναι δύσκολο για μα να αξιολογήσουμε αν κάποια προγράμματα τα οποία ήδη υπάρχουν καλύπτουν κάποιε γραμμέ ή δράσει ή όχι. Γι' αυτό κάναμε αυτή την αξιολόγηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο για να δούμε τι γίνεται σχετικά και αν υπάρχουν κάποιες ε, ελλείψεις ή κάτι το οποίο απουσιάζει, πράγμα το οποίο είναι αναπόφευκτο, διότι υπάρχουν πολλές τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις, καλή ιδέα είναι για κάποια από τα πιλωτικά προγράμματα και υποκατατικές δράσεις που ούτε ή άλλως θα κατατεθούν και για του χρόνου και που θα τα ξαναδούμε, να δούμε αν μπορούν να ενταχθούν ή όχι. Θα σταματήσω εδώ, αυτές οι παρατηρήσεις είχα. Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα, έτσι, ευχαριστώ. Euh, ευχαριστώ και επιμένω σε αυτά που είπε η συγγήτρια όσον αφορά το σχόλιο για τις γραμμές των πιλωτικών προϊόν, προγραμμάτων όπου υπάρχει ήδη ε, δέσμευση των ε, πιστώσεων πληρωμής. Ακόμη λοιπόν και αν ε, υπάρχουν νέα σχόλια για χρήματα όπου υπάρχουν δεσμεύσεις. δεν θα, δεν θα πληρώσουμε κεφάλαια αλλά απλώ θα δεσμευτούμε το οποίο δημοσιονομικά δεν έχει πολύ ε, ε, νόημα. Η Χέλγα, τουλάχιστον θα ήθελα να έχω μια γραπτή δέσμευση, γραπτός μπροστά μου γι' αυτό, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα ληφθεί υπόψη και θα γίνει. Διαφορετικά δεν είμαι πρόθυμη να υπερψηφίσω αυτό το πακέτο προτάσεων. Πρέπει να είναι σαφές με κάποια δέσμευση γραπτός. Διαφορετικά δεν θα το εγκρίνω. Ελγκά, δεν πρόκειται, για, δεν πρόκειται για υπόσχεση, θα το ψηφίσουμε αμέσω. Θα το προσθέσουμε στον πίνακα όπως προσθέσαμε και την ΚΟΥΕ και προσθέσαμε και τους ε, πρασίνους. Πράγμα το οποίο επιτρέπει να ικανοποιήσουμε τις περισσότερες πολιτικές ε, ομάδες που είναι κάτι φυσιολογικό. Εν συντομία. Είχα δηλαδή- υπόψη ότι δεν θα ψηφίζαμε σχόλια σήμερα γιατί είχα αναφέρει ότι θέλαμε ξεχωριστή ψηφοφορία για το θέμα της γραμμής του κονδυλίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία, για αυτή την τροπολογία. Εσείς ζητάτε να υπάρξει την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή χωριστή ψηφοφορία για τις ε, ε, τροπολογίες, για τις παρατηρήσεις. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα είναι όσο αφορά το 363, όπου οι πράσινοι θέλουν να διαγράψουν μια φράση στις παρατηρήσεις. Και εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή τη διαγραφή. Θέλουμε λοιπόν να γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία γι' αυτό, ώστε να μην γίνει αυτή η διαγραφή. Θέλουμε να υπάρξουν αυτές οι παρατηρήσεις. Ωραία, για την επόμενη εβδομάδα λοιπόν. Θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα τις παρατηρήσεις, εντάξει. Τώρα έχουμε μόνο τα ποσά. Κανείς άλλος λοιπόν δεν ζητά το λόγο, οπότε υποβάλλω προς ψηφοφορία τον πίνακα μόνο για τους αριθμούς όλων των ε, ε, προκαταρτικών ε, δράσεων και προσθέτοντας το πιλωτικό πρόγραμμα των Πρασίνων που είναι μέσω συμβιβασμό. Ποιος είναι υπέρ. κατά αποχές μία αποχή. Άρα, ο πίνοκας των πιλωτικών ε, δράσεων έχει ε, ψηφιστεί. Συνάδελφοι, αισθάνομαι ανακούφιση και θέλω να συγχαρούμε θερμά την εισηγήτρια διότι είναι σπάνιο ένα νέο μέλος από την πρώτη χρονιά να αναλάβει την έκθεση και μέχρι στιγμής έχει πάει άψογα και έχω εκτιμήσει όχι μόνο την, ε, ε, ε, την τις ικανότητες τη συντονία με την οποία είχαμε συνεργαστεί στην προηγούμενη τη ζωή ε, αλλά και ε, στην σοβαρότητά της. Ευχαριστώ επίσης διότι όλοι παρίσταντο ίσως κατά καιρού είχαμε και υπερβολικούς εκπροσώπους του ΕΛΚ και δεν μπορούσα να ψηφίσω. μη μου το κάνετε αυτό γιατί μπορεί να αλλάξω κόμμα. Και θέλω να ευχαριστήσω και τους συντονιστές αλλά έχουμε καλύψει μόνο το 1 τρίτον των εργασιών μας. Δηλαδή συμφωνήσαμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, θα ολοκληρώσουμε την επόμενη εβδομάδα, θα επανέλθω σε αυτό, μετά θα συγκαλέσουμε την ε, Ολομέλη για να καταλήξουμε σε μία συμφωνία επί των προτάσεών μας και μετά θα υπάρξει η συνδιαλλαγή. Στη συνδιαλλαγή πρέπει να πούμε ότι για μας τα μέλη της Επιτροπής η διάσκεψη των Προέδρων εν τη σοφία της έχει καταλάβει τα επιχειρήματα που παρουσιάσαμε σχετικά με τη σύσταση της διαπραγματευτικής ομάδας στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής και αντί να ζητήσει ε, να υπάρξει μία στάθμιση ανά επιτροπή αποφάσισε πολιτικά καλύτερα να ακολουθηθεί ο, ο κανόνας de σε κάθε ομάδα. Οπότε Συνάδελφοι, εσείς πρέπει ο καθένας να επηρεάσετε στην πολιτική σας ομάδα του συναδέλφους κατά τρόπον ώστε οι ικανότητες, οι αρμοδιότητες, η ε, εξοικείωση με τα θέματα τα δημοσιονομικά να μπορέσουν να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα στην ε, ε, Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Άρα, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε Δευτέρα και Τρίτη μία συνεδρίαση της ομάδος προπολογισμού για να ψηφίσουμε τα υπόλοιπα ε, δηλαδή τα σχόλια για τις πιλωτικές ενέργειες και τις προκατακτικές ενέργειες ε, όπου οι αριθμοί που πρέπει ακόμη να διευκρινιστούν για να ε, μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την πολιτική συμφωνία στην κατηγορία 4, δηλαδή την κατανομή ε, μεταξύ των ε, γραμμών που αναφέρονται ε, στην μπανάνα και στο ICI Plus και ε, άλλα θέματα όπου ως παραδείγματος χάρη ότι αν έχουμε διακοπή ρεύματος μπορεί να εξαφανιστούν εκατομμύρια ευρώ κάπου θα πρέπει να έχουμε ε, κάποιο απόθεμα, κάποιο buffer, κάποια buffer line για να ξέρουμε ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε ολόκληρη την κατηγορία μας ένα α. Θα ψηφίσουμε επίσης σε μία ή ίσως περισσότερες πολιτικές γραμμές όπως η τροπολογία που κατέθεσαν οι φίλοι σοσιαλιστές για τη δημιουργία ενός νέου πόρου που θα μπορέσει να ε, τροφοδοτήσει τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και αναρωτιόμαστε πώς εμείς θα παρουσιάσουμε τη διαπραγματευτική μας θέση έναντι του Συμβουλίου κατά τρόπον ώστε πέραν του προπολογισμού του 2011 να αρχίσει να σκέφτεται και τη συνέχεια. Δηλαδή πόσο ε, θα ε, εξέλθει από το ε, κυβερνητικό αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Και με αυτό το πνεύμα η διάσκεψη των Προέδρων θα συνέλθει την Τρίτη το πρωί στις 8.30 και εκεί έχω κληθεί με τους δύο εισηγητές κατά τρόπο ώστε να καταρτήσουμε την Ολομέλεια της 20 Οκτωβρίου και τις επιαφές με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι οι ψηφοφορίες οι οποίες προέκυψαν μας δίνουν μία σαφή εντολή για να μιλήσουμε στη διάσκεψη των Προέδρων. Τη Δευτέρα θα διευκρινίσουμε τι ώρα θα ξεκινήσει η Επιτροπή ε, Προϋπολογισμού την Τρίτη το πρωί. Μπορεί να αργήσουμε λιγάκι γιατί αντί ε, για 9 ίσως ξεκινήσουμε 9.30-10 θα πάρει μια ώρα η διάσκεψη των Προέδρων και θα πρέπει επίσης να δούμε εάν τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξει η διάσκεψη των Προέδρων θα μας οδηγήσουν σε μία προσαρμογή του σχεδίου ψηφίσματος που θα ψηφιστεί επίσης στις 20 Οκτωβρίου, διότι Εάν θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στο Συμβούλιο, σε αυτό το επίπεδο, Ίσως δεν θα γίνει ε, συγκεκριμένα για τη γραμμή του προϋπολογισμού αλλά για να θέσουμε ε, τον προϋπολογισμό του 2011 σε μια ευρύτερη ε, προοπτική. Οπότε μια δυνατότητα που έχει το Κοινοβούλιο στα πλαίσια αυτά είναι να εφαρμόσει αυτή την επέκταση στο σχέδιο ψηφίσματος. Για το σχέδιο ψηφίσματος Καταρχήν, θα πρέπει να μας έχουν κατανεμηθεί οι τροπολογίες. Πρώτα θα πρέπει να έχουν κατατεθεί. Υπάρχει μία προθεσμία για τις 4 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι, αλλά καλό θα ήταν ήδη να τα είχαμε στο τέλος αυτής της εβδομάδας, να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε το Σαββατοκύριακο ή τουλάχιστον ε, κάποια προηγευθεί για να ξέρουμε περί τίνος θα ομιλούμε. Μου επιτρέπετε για να αποσαφηνίσω αυτό το θέμα. Έχω αρκετά προχωρήσει στο σχέδιο ψηφίσματος για το ψήφισμα. Ελπίζω να το έχω έτοιμο και να το έχω διατυπώσει, όχι τελεσίδικα, αλλά να το έχω ολοκληρώσει ως σχέδιο σήμερα και να σας έχει διανεμηθεί μέχρι αύριο, ώστε να είναι στη διάθεσή σας. Αύριο θα το έχετε σίγουρα. Καλό θα ήταν να το έχουμε πριν το Σαββατοκύριακο. Εγώ θα δουλέψω το Σαββατοκύριακο, ιδίω ε, όσον αφορά τι λεπτομέρειε των τροπολογιών. Ιάν. Είπατε πολλά ωραία πράγματα στη συντόνια και νομίζω ότι αξίζει. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν εξαιρετική συγγήτρια μέχρι τώρα. Πολλή δουλειά υπάρχει ακόμα βέβαια που πρέπει να κάνει ακόμα. Και εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια επένων προς τον Πρόεδρο, γιατί προεδρεύσατε με πάρα πολύ καλό τρόπο αυτή τη συνεδρίαση. Στη γραμματεία όμως να απευθύνουμε επένους, γιατί χωρίς τη γραμματεία είμαι τίποτα εγώ, δεν καταφέρνω τίποτα. Ναι και στη γραμματεία, σίγουρα, διότι έκανε και η γραμματεία εξαιρετική δουλειά, είναι πάντα πολύ δύσκολο και όταν μάλιστα κόβεται και το ηλεκτρικό ρεύμα και δυσχεραίνεται ακόμα πιο πολύ δουλειά, θα ήθελα να προσθέσω μια μικρή ανησυχία που έχω. Το χαιρετίζω ότι οι ηγέτες αυτού του σώματος έχουν μεγάλο ενδιαφέρον στην ε, δουλειά που κάνει η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ο προϋπολογισμός είναι, ας το πω εσύ, το σημαντικότερος μοχλός των εξουσιών του Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικότατο μέσο λοιπόν. Θα ήθελα απλά και μόνο όμως να πω ότι φαντάζομαι ότι η βασίλισσα της Αγγλίας είναι υπέρ των δικών της κοσμημάτων του στέματος, αλλά δεν τα φυλάει η ίδια, δεν τα φρουρεί η ίδια. Κάποιος ε, ειδικό για την ασφάλεια έχει επιφορτιστεί την ε, φύλαξη των ε, κοσμημάτων του στέματος. Είναι μια πολύ καλή αρχή αυτή και πρέπει να ισχύει και για μας. Merci, Anne, pour cette... Ευχαριστώ αν για αυτή την τελευταία παρατήρηση και για τους επένους. Οπότε αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι πάντοτε όταν το Κοινοβούλιο δουλεύει καλά πρόκειται για συλλογική εργασία και γι' αυτό είμαστε περήφανοι ότι συμμετέχουμε σε ένα έργο που δεν θα αφήσει κανείς μεμονωμένα το όνομά του. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ. Έχουμε τελειώσει μια ώρα πιο πριν. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς. Είναι πάντοτε πολύ δύσκολο να ερμηνεύουμε τις ψηφοφορίες του προϋπολογισμού. Διαβάστε καλά το Σαββατοκύριακο, μελετήστε το σχέδιο ψηφοφορίες και θα σας δίνω ραντεβού τη Δευτέρα, λύεται η συνεδρίαση.